Ε, ελέγχουν τη συζήτηση. Και αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Εάν αυτοί ελέγξουν την κατεύθυνση της συζήτησης, αυτό που ήταν ε, οι ιδεολογίες, ε, ο κομμουνισμός και ο ρατσισμός, που ήταν αυτές οι ακραίες ιδεολογίες, θα αντικασταθούν με τον οικολογισμό και τον καταστροφολογία για το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό κύριο κύριος Κόκαλης. Madam President, Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ε, προώθηση αυτού του θέματος, διαφωνώ με το τίτλο. Είναι επίγουσα κατάσταση. Είναι κάτι το απροσδόκητο, χρειάζεται άμεση δράση. Αλλά δεν είναι κλιματική καταστροφή ή οικολογική καταστροφή. Είναι καταστροφή που προκάλεσαν οι άνθρωποι, που καταστρέφει τις αλυσίδες επισητισμού, δημιουργεί καταστραμμένα κράτη, δημιουργεί κλιματικούς πρόσφυγες, ε, ξεπερνά τις δυνατότητες που έχουμε για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό μας από ακραία καιρικά φαινόμενα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε την επίγουσα αυτή κατάσταση. Η Ευρώπη όμως μπορεί να είναι στην πρωτοπορία στην αντιμετώπιση. Το πρωί είπαμε ότι υπάρχει επίγουσα κατάσταση στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Στην ε, σημερινή όμως, στην τωρινή τώρα συζήτηση, είμαστε ηγέτες στην αντιμετώπιση και θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε. Μέχρι την Άνοιξη αναμένουμε να εγκρίνουμε μια δίκαια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Δηλαδή θα χρειαστούμε μια ε, ολιστική και οριζόντια πλατφόρμα με νομοθεσία και σχέδια δράσης για να έχουμε την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Και παράλληλα θα δημιουργήσουμε και εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και θα εξοικονομήσουμε και 3 εκατομμύρια εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Δεν έχουμε επαρκή στην Ευρώπη. Άρα δεν θα χαθούν θέσει εργασία. Πρέπει να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίγουσα κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Κοράου. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον θεωρητικό θέμα μεταξύ των επιστημόνων. Είναι στη γειτονιά μας. Ε, είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν δράσουμε αποφασιστικά θα υπάρχουν καταστρεπτικές συνέπειες ε, στο παρόν αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά δεν συνδέονται πια με ακραίες ιδεολογίες. Είναι ένα σημαντικό θέμα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος και εμπλέκει όλη την ανθρωπότητα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος για αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να είναι η ξεκάθαρη πρόταση της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς, είναι ουσιαστικό να αφαιρέσουμε τις πληρωμές για το πρασίνισμα από τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και τα κράτη-μέλη δύσκολα μπορούν να δράσουν σωστά. Δεύτερον, πρέπει σταδιακά να, ε, να απομακρυνθούμε από τις επενδύσεις ε, στα ορυκτά καύσιμα. Επίσης, ε, πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση των, των στόχων να έχουμε 65% μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Οι μελλοντικές γενιές θα μας κρίνουν για αυτό που κάνουμε στον πλανήτη και ε, θα είναι σκληρή αυτή η κρίση. Χρειαζόμαστε να αναλάβουμε δράση τώρα. Ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό η κυρία Τότ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, να τονίσω ότι η αναθέρμανση του πλανήτη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε επιγόντως. Υπάρχουν επιστημονικά γεγονότα που, και δεδομένα που μας αποδεικνύουν ότι δεν είναι αργά να επιβραδύνουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να έχουμε καλά ε, καταρτισμένα σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να συνεισφέρει στις δαπάνες των κρατών μελών αν θέλουμε πραγματικά η ευρωπαϊκή οικονομία να είναι ουδέτερη σε επίπεδο εκπομπών μέχρι το 2050. Το 90% της ενέργειας στην Ουγγαρία μπορεί να είναι μέχρι το 2030 ε, ουδέτερο σε επίπεδο εκπομπών. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι το κόστος αυτής της ουδετερότητας μπορεί να φτάσει τα 150 δις ευρώ. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει προτεραιότητα ε, ως προς τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας ε, σε συνδυασμό με την τήρηση των περιβαλλοντικών στόχων. Νομίζω λοιπόν ότι στο μέλλον πρέπει να βρεθεί μία λύση κόστος ε, του να είναι κανείς περιβαλλοντικά ουδέτερος ε, να επιμερίζεται έτσι ώστε οι χώρες της Ευρώπης και η Ευρώπη γενικά να είναι ανταγωνιστικές. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριος Μπόμεν. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, το μήνυμα από, από τη Νέα Υόρκη ήταν ξεκάθαρο. Η Σύνοδος Κορυφής για την Αηφορία ε, ήταν ε, ε σε χαρτί και πραγματικά είμαστε στο σωστό δρόμο, Επίτροπε, όμως ε, τελικά επιστρέφουμε σε αυτά που είχαμε ξεκαθαρίσει και σε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση να πάμε μπροστά και εμείς ε, στα δικά μας πολιτικά πεδία στον εσωτερικό μας προϋπολογισμό να δώσουμε τη νέα κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει και στη μετάβαση προς τη νέα Κομισιόν. Έχει περιγράψει ένα σενάριο η νέα Κομισιόν που θα είναι δεσμευτικό για το περιβάλλον για όλες ε, τις ε, πολιτικές διαστάσεις. Όμως δεν έχω ακούσει κάτι δεσμευτικό αυτή τη στιγμή ακόμα. Ε, αυτό το σενάριο 1 θα είναι, λέει, η πηξίδα της νέας επιτροπής. Ε, θέλουμε όμως αυτό να το δούμε και να το ακούσουμε. Γιατί πραγματικά αυτό θα είναι μεγάλη συμβολή στην ε, μετάβαση προς τη νέα αυτή επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Ρίση έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας είμαστε σαφείς και ειλικρινείς. Η Σύνοδος για την Κλιματική Αλλαγή στην Νέα Υόρκη ε, είχε μόνο 68 χώρε που αντιστοιχούν μόνο στο 7% των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα και ουσιαστικά είχαμε πενιχρά αποτελέσματα. Οι μεγάλοι όμω ε, ρηπαντέ, οι χώρε οι οποίε μολύνουν περισσότερο από όλε τι υπόλοιπε, δεν ήταν παρούσε. Θα πρέπει η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υποδειγματική. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι το Green Deal, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα χίλια δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια τα οποία θα πρέπει να επενδυθούν στην οικολογική μετάβαση με πολύ κεντρικό ρόλο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά φαίνονται ευνόητα, αλλά τη στιγμή που συρρυκνώνονται οι φιλοδοξίε για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο 2021 με 2027, θα πρέπει και τα ευνόητα πράγματα να τα επενθυμίζουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να μειώσουμε την ρήπανση στην ατμόσφαιρα, την ρήπανση που βάλει κατά τη υγεία μα και μην ξεχνάμε ότι είναι ακριβώ η ρήπανση αυτή που ευθύνεται για 670 θανάτους ε, το χρόνο στην ε, Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να αποτελέσει αυτό προτεραιότητα για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώς επειδή οι πολίτε πρέπει να έχουν μια σωστή υγεία μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Χόλμγκρεν τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά αντιμετωπίζουμε μια επίγουσα κατάσταση, μια έκτακτη ανάγκη όταν μιλάμε για την βιοπικιλότητα και όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Η βιοπικιλότητα είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε να προσαρμοστούμε στην κλιματική αλλαγή. Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή την κρίση σαν ήταν πραγματικά κρίση. Περάσαμε το κατώτατο όριο της αύξησης του ενός βαθμού Κελσίου και τα πράγματα επιδεινώνονται. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μειώσει την υπερθέρμανση του πλανήτη μέσω της καλλιέργειας συγκεκριμένων φυτών, συγκεκριμένων δέντρων. Θα μπορούσαμε να είχαμε σημειώσει και επιτυχία με τη Συμφωνία των Παρισίων, αλλά η βασική προπόθεση είναι τα επόμενα πέντε χρόνια να καταβάλουμε άοκνε προσπάθειε. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο κατεβαίνουν οι νέοι στου δρόμου και διαδηλώνουν παντού στον κόσμο. Τα πέντε αυτά χρόνια είναι τα καθοριστικά τελευταία πέντε χρόνια που θα έχουμε στη διάθεσή μα, προκειμένου να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε τον πλανήτη μα στην κλιματική αυτή αλλαγή. Επομένω, θα συσπηρωθούμε και θα συναλάβουμε δράση. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν πρέπει να χαιρόμαστε επειδή όλη η πολιτική κλάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολείται πλέον με την οικολογία, από την άλλη υπάρχει μια έντονη ιδιοτέλεια και κεροσκοπία την οποία την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο του greenwashing, όπου προσπαθούμε ουσιαστικά να προσδώσουμε μια οικολογική έκφανση σε πάρα πολλέ πολιτικέ που ακολουθούμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πάρα πολλά κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ουσιαστικά δεν ακολουθούν μια οικολογική πολιτική, αλλά έχουν ε, τεθεί σε ένα είδο φορολογική ομοιρία εξαιτία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνουμε τις ευθύνε στου πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δι στους πιο άπερου πολίτες, ενώ θα έπρεπε να καταδικάσουμε ουσιαστικά τις εθνικές πολιτικές που ακολουθούνται. Νομίζω ότι είναι η ίδια η οικονομική πολιτική, η ιδεολογία η οποία πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου πραγματικά να τα αποκριθούμε στην περιβαλλοντική και ηθική, θα έλεγα, διοντολογική αυτή έκτακτη ανάγκη. Όλα έχουν να κάνουν με τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών και έχουν να κάνουν επίση και με την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτά είναι βασικέ προποθέσει. Όλα τα υπόλοιπα είναι περί τα λόγια. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Βυσνιέσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ακούω εδώ τη συζήτηση. Αλλά δεν άκουσα ούτε λέξη για τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα του συστήματος ETS, εμπορίας εκπομπών. Ούτε άκουσα τίποτα από την αριστερή πλευρά για την ενεργειακή παινία. 55 εκατομμύρια συμπολίτες μας ε, την υφίστανται. Και τι θέλετε σήμερα. Θέλετε να καλύψετε με τις περιοριστικές πολιτικές σας και άλλους τομείς. Για παράδειγμα τη γεωργία θέλετε να επεκταθεί και εκεί η ενεργειακή παινία. Ωραία. Ξέρετε, εκτός Ευρώπης θα μεταφερθεί τελικά η γεωρική παραγωγή. Με αντιβιωτικά, με ό,τι θέλετε. Άρα χρειαζόμαστε μια πολιτική που να είναι λογική και ισορροπημένη. Που να επιτρέπει να αναπτυχθούν τα κράτη-μέλη μας, να αναπτύσσει η οικονομία μας. Και που δέχεται το δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους μείγμα. Μια τέτοια πολιτική θα επιτρέπει να αναπτυσσόμεθα όλοι όπως μπορούμε για να μειώσουμε τελικά και την ενεργειακή φτώχεια. Ευχαριστώ ε, ο κύριος Βουάλλας. Στη συνάντηση κορυφής συζήτησαν 10 λεπτά την κλιματική δράση. Ε, αυτό δείχνει που είναι η προτεραιότητά τους. Στη συνάντηση στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα υποτίθεται ότι θα κάναμε περισσότερα. Και τελικά μου όρος και οι επιστήμονες το καθιστούν σαφές. Κανένας από του στόχους μας δεν συμβαδίζει με τους στόχους των Παρισιών. Ούτε για το κλίμα, ούτε για την ε, ενεργειακή κατανάλωση. Η κατάσταση επίγουσα χρειάζεται και επίγουσα αντίδραση. Αν θέλετε σοβαρά να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα του κλίματο. πρέπει να κάνουμε ορισμένα πράγματα τώρα. Πρέπει να σταματήσουν τώρα οι επιδοτήσει στα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να σταματήσουν τα προγράμματα για υγροποιημένο φυσικό αέριο παντού στην Ευρώπη και αυτό στο Σάνον. Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται το φυσικό αέριο και θα πρέπει να σταματήσει να ισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, αρνούμαστε την πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ενάμιση λεπτό. Ο κύριος Λίντς. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα που προκαλεί έντονα συναισθήματα. Το είδαμε και στις ε, διαδηλώσεις των μαθητών που γίνονται κάθε Παρασκευή. Και εδώ όμως σήμερα ήταν σαφές. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνουμε. Είναι ότι ορισμένοι αγνοούν την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να δαιμονοποιούμε ορισμένους κλάδους της οικονομίας. Πρέπει να τονίσουμε ότι μπορούμε να λάβουμε θετικά μέτρα. Μόνο εάν τα μέτρα τα δέχεται η κοινωνία θα επιτύχουν. Ένα παράδειγμα από τη Γεωργία. Οι Γεωργοί ζορίζονται γιατί πάντα κατηγορούνται αυτοί ότι καταστρέφουν το κλίμα παντού στην Ευρώπη. Και διαδηλώνουν. Χθε και εδώ, μπροστά στο Κοινοβούλιο. Γιατί ξεχνάμε στη συζήτηση ότι η γεωργία και η δασοκομεία είναι οι μόνοι τομεί που έχουν τεράστιες δυνατότητες δέσμευση διοξιδίου του άνθρακο. Τα δάση μας δεσμεύουν τουλάχιστον 10% από τις εκπομπές μας. Γι' αυτό αντί για την ε, αποφυγή παραγωγής θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με τη δέσμευση. Τέτοιοι μηχανισμοί κινήτρων θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Για παράδειγμα η Νέα Ζηλανδία έχει ε, ακολουθήσει αυτήν την οδό. Παρακαλά, παρακαλώ να, επενε, ε, να επενούμε τους γεωργούς μας για αυτά που κάνουν και όχι να τους κατηγορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ. Η αντίπετ... Τόπιση της έκτακτης ανάγκης ε, στο κλίμα πρέπει να είναι το καθοριστικό θέμα στην Ευρώπη. Οι ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, μεταφορές, ωκεανοί, η ε, ε, συμφωνίες συναλλαγών ε, που προστατεύουν το κλίμα, ψηφιοποίηση, περιφερειακή ανάπτυξη, αηφόρο επένδυση. Όλα αυτά θα πρέπει να αγκαλιάζουν τους ενδιαφερόμενους, τους εμπειρογνώμονε και τους πολίτες. Ε, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία η οποία ηγείται στον κόσμο θα είναι στο, και θα πρέπει να είναι στο χαρτοφυλάκιο κάθε επιτρόπου και κάθε ευρωπαϊκής κυβέρνησης. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα καταστροφικό χάος αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβει άμεση και ολιστική δράση. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση είμαστε οι, Ευρωπαίοι πολίτες ε, σε... μια κατάσταση που δεν πρέπει κανείς να μείνει πίσω. Ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι γυναίκες, ούτε κανένας πολίτης. Ο αέρας που αναπνέουμε πρέπει να παραμείνει καθαρός για τους νέους. Ε, δεν πρέπει να περιμένουμε ούτε μία στιγμή. Πρέπει αυτή τη στιγμή να κηρύξουμε έκτακτη ανάγκη σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όντως έχουμε μια εκτακτή ανάγκη, αλλά δεν πράττουμε σαν να είμαστε σε εκτακτή ανάγκη. Δεν είναι ότι ε, δεν το ξέρουμε, το αγνοούσαμε τόσο καιρό και τώρα έφτασε στην πόρτα μας. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι... Ε, ότι πρέπει να αντισταθούμε για να προστατεύσουμε τις μέλισσες, την βιοπικιλότητα, ε, να αντισταθούμε. Ε, φέτος ε, εκλεγήκαμε με την εντολή, την ισχυρή εντολή να δράσουμε στο κλίμα και στη βιοπικιλότητα. Τι πρέπει τώρα να κάνουμε λοιπόν, να κάνουμε τα κράτη, τις κυβερνήσεις να λογοδοτήσουν. Γιατί ναι, μπορεί σταδιακά να φεύγουμε από τον άνθρακα, αλλά δίνουμε χρήματα για εργοστάσεις για παραγωγή ηλεκτρισμού. Λέμε να πάμε στις ανανεώσιμες και ταυτόχρονα έχουμε ε, αγωγούς ε, πετρελαίου που χτίζονται με κοινό συμφέρον όλων. Έτσι λοιπόν πρέπει όλες οι κυβερνήσεις να λογοδοτούν και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Αντελή. Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε το πιο θερμό έτος. Ε, η έκτακτη ανάγκη στο κλίμα είναι κάτι που ζούμε κάθε μέρα. Ήδη πλήττει τους πληθυσμούς που είναι οι πιο ευάλωτοι. Τέλειωσε ο χρόνος των διασκέψεων και των συζητήσεων. Ε, πρέπει να διαπιστώσουμε. Με λείπει ότι πρέπει με ε, άμεσα να αντιδράσουμε σε αυτή την έκτακτη ανάγκη με δράση. Εμείς πρέπει καταρχάς να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να, να μειώσουμε τις εκπομπές μας μέχρι το 2030 ώστε η ναυτιλία, η αεροπλοεία ε, να πληρώνουν φόρους και να συμμετάσχουν σε αυτή τη μετάβαση. Είναι η μάχη του κλίματος, της εργασίας, ε, της ευημερία, ε, η κοινή μας μάχη, αυτή που δίνουμε όλοι οι πολίτες ε, και αυτό που πρέπει να δείξουμε σε αυτή την νεολαία που έχει βγει στους δρόμους, που μας κοιτάει στα μάτια, που περιμένει από μας. Πρέπει να τους δείξουμε ότι τελικά έχουμε καταλάβει το μήνυμα και ότι έχουμε το πολιτικό θάρρος να πούμε ξεκάθαρα και σωστά ότι θα είμαστε γρήγοροι, ισχυροί και σωστοί σε αυτά που κάνουμε. Για ένα λεπτό ο κύριος Λαντσίνη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι πρόσφατε διαδηλώσει για την κλιματική αλλαγή που προβλήθηκαν πάρα πολύ από τα μέσα ενημέρωση παρουσίασαν καταστροφικά σενάρια χωρί να παρέχουν πραγματικέ λύσει. Η Ευρώπη έχει ήδη μειώσει πάρα πολύ τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα η Γαλλία μα προτείνει να πετύχουμε τη λεγόμενη κλιματική ουδετερότητα ήδη μέχρι το 2050. Ένα αξιέπαινο στόχο, ο οποίο θα είναι ιδιαίτερα ευνίδιο και, αξι... και επιζήμιο όμω για του πολίτε και τι επιχειρήσει μα. Η Ιταλία, έχοντα κάνει πάρα πολλέ επενδύσει, θα πετύχει ήδη μέχρι το 2020 την κατάργηση τη χρήση άνθρακα. Άλλε χώρε όμω, οι οποίε δεσμεύονται από το Σύμφωνο Σταθερότητα, εξακολουθούν και χρησιμοποιούν άνθρακα ή ακόμα και για το 40% του ενεργειακού τους μείγματος. Και βέβαια οι χώρες αυτές δεν μπορούν να φτάσουν τους στόχους αυτούς. Είναι λοιπόν πιο σημαντικό να τηρούμε του εσκαλισμένου προπολογισμού ή την προστασία του περιβάλλοντο. Και όποιο δεν τηρεί τι παραμέτρου στην περίπτωση αυτή δεν θα καταβάλει το τίμημα. Ξέρετε ότι η ρήπα δεν σταματάει στα εθνικά σύνορα. Συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίε με χώρε οι οποίε δεν έχουν περιβαλλοντικέ δεσμεύσει και υποχρεώσει. Εισάγουμε τα προϊόντα του, συμβάλλουμε κατά αυτόν τον τρόπο και εμεί την ρήπανση και δημιουργούμε αθέμητο ανταγωνισμό ει βάρο των δικών μα των επιχειρήσεων, οι οποίε δικαιολογημένα υπόκεινται σε πολύ αυστηρού περιβαλλοντικού κανόνε έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα χαντάκι και προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει από αυτό σκάβοντας όλο και πιο βαθιά. Σας ευχαριστούμε κυρία Κλόκτστορ. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευθύ αμέσω πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος ορισμός για την κλιματική απειλή Εκτιμώ τις ανησυχίες που έχετε για το μέλλον, για το περιβάλλον μας και που ενδιαφέρεστε για όλες αυτές τις βασικότατες ανθρώπινες αξίες. Τι θα πει όμως κλιματική αλλαγή, κλιματική καταστροφή. Βλέπουμε ότι το κίνημα Extinction Rebellion μας προβάλλει διάφορα βίντεο, διάφορες ταινίε που έχουν δημιουργήσει προκειμένου να μας ανησυχήσουν ακόμα περισσότερο. Έχω την εντύπωση όμω ότι δεν γνωρίζουν τελικά και οι ίδιοι τι κάνουν. Χειραγωγούνται, θεωρώ, μόνο και μόνο για να διαχέουν ένα καθεστώ αναρχία. Αυτό είναι επικίνδυνο και επίση ανεύθυνο. Η ε, αλήθεια είναι ότι μόνο οι πιο πλούσιοι τελικά και ευκατάστατοι μπορούν να αναλούν το χρόνο τους έτσι διαδηλώνοντας για το περιβάλλον. Και ας μην ξεχνάμε όμως ότι το πραγματικό τίμημα το πληρώνουν οι φτωχοί, οι πιο άποροι, αυτοί ουσιαστικά που υποφέρουν από τη λεγόμενη ενεργειακή ένδυα. Και μου κάνει εντύπωση που έρχεται και το χάβι τώρα όλο αυτό το σενάριο του Extinction Rebellion, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τιμή της ενέργειας, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας τα διάφορα μαρξιστικά εγχειρήματα στο παρελθόν έχουν φέρει μόνο οδύνη και φτώχεια. Α μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, γιατί πολύ φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο κάνουμε τώρα. Η κυρία Πιετικάνεν τώρα έχει το λόγο. Η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει μια προσέγγιση που να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά το μετριασμό και την προσαρμογή τη κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση όλων των άλλων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Όλοι οι πολιτικοί κανονισμοί και όλε οι πολιτικέ πρωτοβουλίε θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει Τη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα επόμενα 30 χρόνια. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν πετυχαίνουμε τα επαρκή αποτελέσματα. Υπολοιπόμαθαν των στόχων που έχουμε θέσει. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε καταρχά τι μελλοντικέ προκλήσει και στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις υφιστάμενες προσπάθειές μας αν πραγματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις αυτές. Χρειαζόμαστε επίσης μια δέσμη για την κυρική οικονομία, χρειαζόμαστε επίσης μια βιώσιμη χρηματοδότηση των πολιτικών μας, τις απαραίτητες επίσης περιβαλλοντικές αξιολογήσεις. Διαφορετικά θα καταβάλουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό τίμημα, το τίμημα της μη ανάληψης δράσης. Ας μην πειθόμαστε αυτή τη στιγμή από τα διάφορα καταστροφικά σενάρια τα οποία μας παρουσιάζουν. Ας αντιμετωπίσουμε τα πράγματα ορθολογικά και ας καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση για τα μελλοντικά μας προγράμματα. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λόπες τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι η κλιματική αλλαγή έχει γίνει πραγματικότητα. Πήγουσα κατάσταση τώρα. Οι επιστήμονες μας το λένε. Αν δεν δράσουμε τώρα, η ζημιά θα είναι ανεπανόρθωτη. Και είναι πράγμα, πράγματι απειλή για τον τρόπο ζωή μας. Το λένε κάθε Παρασκευή οι νέοι όταν διαδηλώνουν για να ζητήσουν ε, αποφασιστική δράση. Μα το λένε τα Ηνωμένα Έθνη που οργανώνουν ε, συναντήσει κορυφή για να ξυπνήσει η διεθνή κοινότητα. Πρέπει να δράσουμε με ευφυή τρόπο, φιλόδοξο και δίκαιο για να μην παράγουμε πλέον ε, οξύδια του, οξυγο, ε, του άνθρακα και να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι το 2050. Πρέπει να δράσουμε στην ενέργεια, στις υποδομές, μέσω φόρων, για τις μεταφορές, το διεθνές εμπόριο. Όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν, κινητοποιώντας επαρκείς πόρους για να γίνει πραγματικότητα αυτή η αλλαγή χρειάζεται μια ευρωπαϊκή νέα συμφωνία και για να υπάρξουν και ε, κοινωνικοί απορροφητήρες κράτασμών. Να το κάνουμε λοιπόν με ευρωπαϊκό τρόπο που είναι ο καλύτερος γιατί δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε το κλίμα. για το κλίμα πρέπει να συνεργαστούμε. Και αυτό προτείνουμε εμείς ως σώμα. Και αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόντεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η σχέση μεταξύ της ανθρωπότητας ε, και της γης που κατοικούμε είναι σε κρίση. Παντού βλέπουμε ε, την απογοήτευση του κόσμου. Τους τελευταίους μήνες 6 εκατομμύρια πολίτες διαδήλωσαν παντού στον κόσμο για να ζητήσουν νομοθέτες να ακούσουμε και να δράσουμε για την κλιματική επίγουσα κατάσταση και να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Πρέπει να τους ακούσουμε. Η φύση δεν χρειάζεται του ανθρώπου, αλλά εμεί τη χρειαζόμαστε. Το πώ θα δράσουμε τώρα και οι επιλογέ που θα κάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντό μα θα καθορίσουν το μέλλον του ανθρωπίνου είδου ε, για τα επόμενα 10.000 χρόνια. Πρέπει να έχουμε ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πρέπει οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νομοθετήματα του επόμενου μήνε να αντανακλούν την οικολογική επίγουσα κατάσταση και το κλιματικό χάος που θα κλειοδοτήσουμε στα παιδιά, τα εγγόνια μας και τις επόμενες γενιές. Δεν είναι δυνατόν να τους ε, απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό κυρία Πάουλους. Το 2009 το κέντρο ανθεκτικότητας της Στοχόλμης δημοσίευσε μία μελέτη όπου παρουσίαζε εννέα πλανητικές οριακές τιμές που δεν πρέπει να υπερβληθούν αν ο πλανήτης είναι να παραμείνει κατοικίσιμος από το ανθρώπινο είδο. είδος. Έχουμε δίκιο που μιλάμε για κρίση για το κλίμα, αλλά υπάρχουν δύο ανώτατα όρια που ήδη τα έχουμε υπερβεί κατά πολλού. Είναι η ακαιρεότητα της ε, βιοπικιλότητας και οι ροές χημικών. Δηλαδή ε, διαλυτό άζωτο και φόσφορος που εισάγονται συνεχώς στο περιβάλλον. Γι' αυτό εξαλείφονται τα είδη ε, σε ταχύτατους και ανεπανάληπτους ρυθμούς. Τι κάνουμε λοιπόν. Την ίδια τη βάση της επιβίωσής μας ε, την υπονομεύουμε. Την βιοσφαίρα που μας δίνει. Πόσμο νερό, έφορα εδάφη και καθαρό αέρα. Περιμένουμε λοιπόν η νέα επιτροπή να υποβάλει ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα δράσης για τη γεωργία, για τη χρήση της γης, για τους ωκεανούς. Αυτό πρέπει να είναι τμήμα της Πράσινης Συμφωνίας, γιατί αλλιώς δεν θα υπερβούμε αυτή την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρος. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή σαν να ήταν ε, ε, το τέλος ε, της εποχής και η καταστροφή του κόσμου. Ο Πλουτών είναι ένα σημαντικό μόριο στη ζωή του πλανήτη. Ο πλανήτης υπάρχει εδώ και εκατομμύρια χρόνια και οι μετρήσεις ε, για το κλίμα είναι τελείως διαφορετικές από τα μοντέλα για την, για την κλιματική αλλαγή. Ε, έχει αλλάξει τελείως διαφορετικά το κλίμα από ό,τι περιμέναμε και είχαμε προβλέψει. Έχουμε περισσότερους τυφώνες ε, και πλημμύρες και ξηρασίες. Βέβαια το επίπεδο της θάλασσας ε, ανυψώθηκε μόνο 1,8 χιλιοστά τα τελευταία 150 χρόνια. Ε, όχι ε, όσο περιμέναμε. Ναι, λιώνουν οι πάγοι στους πόλους, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο περιμέναμε. Πριν από, ε, ε, λίγα, από κάποια εκατοντάδες χρόνια έληξε η εποχή των παγετώνων και δεν είναι περίεργο που τώρα έχουμε την αναθέρμανση του πλανήτη η κυρία Σουίτσα για ένα λεπτό. Οι παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές είναι προφανείς και είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά στο γεγονός ότι χάνουμε τους πάγους, ότι καίγεται ο Αμαζόνιος. Φέτος το καλοκαίρι είδαμε ακριβώς ε, πώς ε, οι θερμοκρασίες έφτασαν στα ύψη. Είχαμε τις πιο ψηλές θερμοκρασίες ε, τον Ιούλιο. Το 2019 θα είναι ένα από τα πιο θερμά έτη, τα πέντε πιο θερμά έτη. Τόσα συμβαίνουν γύρω μας λοιπόν. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, πρέπει να δράσουμε. Και συμφωνώ μαζί σας, εντάξει δεν είναι το τέλος του κόσμου, αλλά είναι έκτακτη ανάγκη. Και είναι σημαντικό που σήμερα συζητάμε το θέμα αυτό. Ε, στην αρχή αυτής της ε, θητείας, στην αρχή της δουλειάς της νέας Κομισιόν. Θα είμαι μέλος αυτής ε, ε, της προσπάθειας και χαίρομαι που η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν έβαλε την Πράσινη Συμφωνία στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ε, και που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τις πρώτες 100 ημέρες. Επίσης χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής μίλησε για μια ειρηνική μετάβαση, μια πράσινη μετάβαση και ε, μίλησε για τη διασφάλιση της εφαρμογής της Συμφωνίας των Παρισίων. Κάποιος είπε ότι η συνάντηση στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβρη δεν ήταν επιτυχημένη. Ναι, αλλά αυτό ήταν μία από τις πρώτες συζητήσεις και πρω... τις πρώτες συναντήσεις μετά τη Συμφωνία των Παρισίων. Πρέπει πραγματικά να δώσουμε μια... αυτό τον πλανήτη στις μελλοντικέ γενιές σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι το βρήκαμε. Αυτό είναι το... Ε, ηθικό μας καθήκον. Ευχαριστούμε. Επόμενη ε, ομιλήτρια η Κατρίν Φαμπρέντ. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι φύση αισιόδοξη. Επομένως θα ήθελα ένα αισιόδοξο μήνυμα να σας στείλω όσον αφορά ένα ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο και ιδιαίτερα πολύπλοκο και αναφέραμε βέβαια στην κλιματική αλλαγή. Μολονότι Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που παρεμποδίζουν την νομοθετική διαδικασία για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής στο Συμβούλιο. Εγώ ελπίζω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει μια νέα πνοή στο εγχείρημα αυτό και είμαι πεπισμένη ότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καταβάλει προσπάθειε προκειμένου να σταθεί στο ύψο των φιλόδοξων στόχων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χρονικό ορίζοντα το 2020 και το 2030. Αλλά α μην είμαστε αφελεί. Αν πραγματικά θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε υψηλού στόχου, θα πρέπει να δώσουμε και τα απαραίτητα μέσα στη βιομηχανία μα, στι επιχειρήσει μα, για να επιβιώσουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό κόσμο. Χρειαζόμαστε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή χρειαζόμαστε φορολογία του διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύει ότι η αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει και θα πρέπει να προστατεύουμε τι επιχειρήσει μα. Ο κύριο Τσέκ έχει το λόγο. Κυρία Τσέκ, με συγχωρείτε. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. α ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι επιστήμονες. Λίγα χρόνια μα απομένουν μόνο προκειμένου να λάβουμε ουσιαστική δράση κατά τη κλιματική καταστροφή. Δεν πρόκειται για μια ακραία στάση, είναι γεγονό. Έρχομαι από ένα κράτο μέλο, στο οποίο έχουμε κάποιε από τι πιο φτωχέ περιφέρειες Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να πω ότι η καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης θα πρέπει να συμβαδίζει με την καταπολέμηση τη φτώχεια, γιατί οι πιο φτωχέ αυτέ περιοχέ είναι και πιο ευάλωτες στις κλιματικού κινδύνου. Και είναι οι αυτέ που έχουν τα λιγότερα μέσα για να καταπολεμήσουν την κλιματική αυτή, αλλά και βρίσκονται στην αφάβλο κύκλο και πρέπει να λάβουμε δράση. Αν η κλιματική λοιπόν αλλαγή απειλεί το βιό και τη ζωή των πιο ευάλωτων ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι η ζωή του δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο, μόνο μία δίκαιη οικολογική μετάβαση μπορεί να μα βοηθήσει να κινηθούμε προ μία φιλοπεριβαλλοντική πολιτική, προ μία κυκλική οικονομία ο νέος επικεφαλής της, του Δήμου της Βουδαπέστης πραγματικά προωθεί αυτή τη στιγμή μια ιδιαίτερα φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Και επίσης συμφωνώ με τις δηλώσεις που έχει κάνει η νέα Πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Φόντε Λάιεν. Χρειαζόμαστε όμω περισσότερη ελεγγύη στα πλαίσια τη περιφερειακή πολιτική. Α μην αφήσουμε πίσω και εκτό κανέναν Ευρωπαίο. Ο κύριο Καγάιμ τώρα έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και πολύ καιρό συζητάμε και κάνουμε δηλώσει για την κλιματική αλλαγή και τα όσα λέμε μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ του. Όταν όμω πρέπει να ψηφίσουμε για άλλε εμπορικέ συμφωνίε, για ενεργειακά προγράμματα τα οποία σέβονται το περιβάλλον, για μια κοινή γεωργική πολιτική, τότε ξαφνικά αλλάζουμε στάση και υπάρχει μεγαλύτερη απόκληση ανάμεσα στα λόγια και στι πράξει. Αυτό και στη Γαλλία, η οποία προωθεί όλα τα επιτεύγματά τη, όπω η Συμφωνία των Παρισίων, αλλά η ίδια σε εθνικό επίπεδο δεν καταφέρνει τελικά να προωθήσει συγκεκριμένου στόχου Γι' αυτό το λόγο προσέφηγαν κατά τη γαλλική κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στο Ανζόν, την πόλη όπου ήμουν δήμαρχο για πάρα πολύ καιρό. Όπου βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα που λόγω τη κλιματική αλλαγή θα χρειαστεί να εκτοπιστεί σε μια άλλη περιοχή τη Γαλλία στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα να αναλάβουμε δράση. Αυτή τη στιγμή κάνουμε δηλώσει για την οικολογική έκτακτη ανάγκη, αλλά θα πρέπει, πιστεύω, πέρα από τι δηλώσει αυτέ, να καταλήξουμε σε ένα δεσμευτικό νομοθετικό κείμενο. Αν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένε δεσμεύσει και υποχρεώσει για τον προπολογισμό, μπορούμε να έχουμε κάτι τέτοιο για το περιβάλλον και για το κλίμα. Οι υποχρεώσει αυτέ θα πρέπει επίση να είναι και κοινωνικέ, γιατί οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε πέρα από κλιματικέ είναι και κοινωνικέ. Ο συνάδελφο Φανόβερτ, θέλετε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι σημαντικότατη πρόκληση. Για μένα είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ανάπτυξη και μια κυκλική οικονομία. Αυτή θα πρέπει να είναι βασική μας στόχη μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και μέσω της καινοτομία. Το θέμα δεν είναι να καταφέρουμε απλώς να έχουμε ως στόχο το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προστασία του πλανήτη γενικά και αόριστα, θα πρέπει και η πολιτική μας οικονομική και η πολιτική απασχόλησης και η κοινωνική μας πολιτική να διέπεται από περιβαλλοντικούς κλιματικούς στόχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ουσιαστικά να διέπεται από μια οικολογική βιωσιμότητα η ίδια οικονομική μας ανάπτυξη. Πρέπει να βασιστούμε επίσης και σε νέες καινοτόμε λύσεις. Και σίγουρα δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα αυτά μόνοι μας, χρειαζόμαστε και κέριους συμμάχους. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει και απευθύνομαι τώρα στον Επίτροπο. Ποια είναι η στόχη σας προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να συνδέσουμε περισσότερο την πολιτική μας με την πολιτική άλλων τρίτων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και έχει να παρουσιάσει φιλόδοξους στόχους όπως η κατελάχιστον μείωση κατά 50% των εκπομπών του διοξυδίου του άνθρακα έως το 2030. Είναι όμως απαραίτητο να προχωρήσουμε σε μελέτη επιπτώσεων ώστε να μπορούμε να κάνουμε τις υποσχέσεις πράξη και συγχρόνως να παρακολουθήσουμε από κοντά την εφαρμογή των μοντέλων της κυκλικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε όμως επίσης και τους υπόλοιπους παγκόσμιους παίκτες σε αυτή την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όχι μόνο τα κράτη αλλά και πολιτείες και περιφέρειες και περιοχές και οργανώσεις πολιτών. χρειαζόμαστε επίσης και βιώσιμη χρηματοδότηση. η ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων μπορεί να εξελιχθεί σε τράπεζα για το κλίμα είναι όμως απαραίτητο να δώσει την ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης συνεχίζοντας τη χρηματοδότηση των υποδομών του φυσικού αερίου επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει έμπρακτη στήριξη στα κράτη μέλη τα οποία βάζουν φιλόδοξους στόχους στόχους για την ενεργειακή μετάβαση. η χώρα μου η ελλάδα πρόκειται να μειώσει το αποτύπωμα του άνθρακα και να το μηδενίσει το. 2028. είναι λοιπόν απαραίτητο μέσα σε αυτή την προσπάθεια να υπάρξει και η ανάλογη στήριξη. σας ευχαριστώ πολύ. Είχα 1,5 λεπτό, λέει η κυρία Σπυράκη. Μα εγώ έχω ένα λεπτό, λέει η πρόεδρο. Για τους υπόλοιπου ομιλητέ, πάντα ένα λεπτό. Δεν θα το λέω συνέχεια για τον καθένα. Τώρα λοιπόν ο συνάδελφο Μπέλκα. Ευχαριστώ πολύ. Η μετάβαση από την, ε, τα ορυκτά κάψιμα στην παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα έχει μεγάλο κόστος και κοινωνικό, μεγαλύτερο σε ορισμένες χώρες από άλλες. Στην Πολωνία έχουμε μια ακραία περίπτωση, πολύ ψηλό κόστος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνει, γιατί είναι προς το συμφέρον και της ίδιας της χώρας και του περιβάλλοντός της. Διότι λόγω του άνθρακα και ο αέρας μας και τα ύδατά μας είναι μολυσμένα. Η Πολωνία θέλει περισσότερο χρόνο και περισσότερη χρηματοδότηση. Λογικό είναι αλλά μόνο αν οι πολωνικές αρχές δείξουν αποφασιστικότητα για να αλλάξουν το ενεργειακό μείγμα από τα ορυκτά στις ανανεώσιμες. Και περισσότερο χρόνο. Αλλά ναι, η κυβέρνηση πρέπει να παρουσιάσει ένα αναλυτικό, αξιόπιστο, επαληθεύσιμο και αυστηρά παρακολουθήσιμο πρόγραμμα για να περάσει από τα ορυκτά στις ανανεώσιμες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σαν Φλέγκο. Ευχαριστώ πολύ. Το κλίμα και η οικολογία δεν είναι μόνο θέματα μέλλοντος, αλλά παρόντος. Αυτά που συμβαίνουν με το κλίμα, με τις πλημμύρες, με τις ξηρασίες, δεν είναι τυχαία. Και γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουμε επιγόντως. Πρέπει να έχουμε ένα πράσινο βιώσιμο πρόγραμμα, κοινό. Χρειαζόμαστε μια νέα Ευρώπη. Μια Ευρώπη που να μπορεί να συνδυάσει από τη μία την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης με από την άλλη πλευρά μια ε, οικονομία που να αναπτύσσεται και να παράγει ευημερία. Συνάδελφοι, πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ που υπάρχουν προτάσεις για να γίνει μια δίκαιη μετάβαση μέσω του προπολογισμού. Αυτό θα γίνει μόνο ε, εάν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο στραφεί προς την οικολογία. Θέλουμε εναλλακτικέ ε, πηγές ενέργειας. Νέα αυτοκίνητα, καθαρά, αλλά δεν πρέπει να το πληρώσουν οι συμπολίτε μα αυτό. Ο προπολογισμό πρέπει να βοηθήσει. Μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Ανιές. Ε, ο συνάδελφο Κουφ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα επιτύχει μόνο εάν πραγματικά αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Στις μεταφορές και στο περιβάλλον αντιμετωπίζουμε προκλήσει. Ο Φραν Τίμερμαν και ο Κάντρι Σίμψον έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Το αστικό θεματολόγιο είναι ένα καλό σημείο αφετηρίας. Διότι θέτει την στέγαση, την αστική φτώχεια και την ποιότητα του αέρα στη καρδιά μιας δίκαιης μετάβασης μέσω σωστών κανόνων χρηματοδότησης και γνώσης. Κύριε Τίμερμανς, θέλω να ενθαρρύνετε το, την ενεργή ε, τις ενεργείς συγκοινωνίες, δηλαδή να πηγαίνει στη δουλειά του με το ποδήλατο ή περπατώντας. Και η πολεοδομία πρέπει να συνδυαστεί με τις πολιτικές μεταφορών, ούτω ώστε να χρειάζεται να μετακινούνται λιγότερο και ευκολότερα οι άτομοι. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, ε, μόνωσης και του σωστού ενεργειακού εξοπλισμού των κατοικιών για να παράγουμε περισσότερη πράσινη ενέργεια που να πηγαίνει εκεί που χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Ευρέν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πόλεις είναι υπεύθυνε για το 70% των εκπομπών διεξιδίου του άνθρακα. Παίζουν έναν στρατηγικό ρόλο στη μάχη κατά της θέρμανσης του κλίματος. Είμαι κατηγορηματική κύριε Επίτροπε. Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκτακτή ανάγκη στο κλίμα αν δεν μιλήσουμε για τις πόλεις. Η διαπίστωση είναι πολύ απλή. Πολύ συχνά οι πόλεις και μεταξύ αυτών οι μετροπόλεις, μητροπόλεις ξεχνιούνται στη συζήτηση. Και εδώ δεν κάνουμε εξαίρεση. Στο Παρίσι το ξαναβλέπω κάθε μέρα. Οι μητροπολιτικές περιοχές ασφικτιούν μαζί και οι πολίτες. Χάνονται το, χάνεται το πράσινο. Γενικά όλα αυτά ευθύνονται για την ε, θέρμανση του πλανήτη. Πρέπει πραγματικά να δούμε πώς αυτά συμβάλλουν και στην επιδείνωση της υγείας των πολιτών. Αυτά είναι κομμάτι του προβλήματος αλλά και της λύσης, γιατί υπάρχουν πολλές καινοτόμες πρωτοβουλίες που είναι αποτελεσματικές. σας. βάλουμε λοιπόν στην Πράσινη Συμφωνία της πόλης ε, στην καρδιά της συμφωνίας αν θέλουμε επιτυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, Λαλούκ, έχει το λόγο η επόμενη συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για την συζήτηση αυτή. Όντως υπάρχει μια εκτακτή ανάγκη και μια νέα πράσινη συμφωνία. Είναι μια νέα συμφωνία η οποία θα μας μας έφτασε ε, στον τοίχο και τώρα έχουμε μιλήσει ε, πια για την αλλαγή του κλίματος. Είναι ένα σχέδιο για όλη την κοινωνία, ένα σχέδιο για επενδύσεις μαζικό στις low-tech και όχι στις high-tech, στις ε, υποδομές της φυτικής Γενικά σε οποιαδήποτε τομέα μας βοηθά να μειώσουμε τις κλιματικές αλλαγές, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, να φτιάξουμε μια βιομηχανική πολιτική για την Ευρώπη. Θα είναι δύσκολο γιατί όλοι κολυμπάμε στη μαζική κατανάλωση, όμως το, ο ρίσκο είναι να μην είμαστε φιλόδοξοι, είμαστε σε μια ε, κατάσταση επικίνδυνη. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους. Ε, φανταστείτε τι θα γίνει με τους κλιματικούς πρόσφυγες. Ας είμαστε στο ύψος των περιστάσεων σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, Επόμενος, ο, η επόμενη συνάδελφος Βιλμπάου Αράντικα. Οι αλλαγέ που γίνονται στο περιβάλλον από τη δράση του ανθρώπου κάνουν τα ακραία φαινόμενα όλο και πιο συχνά. Θα έχουμε κλιματικέ ε, μεταναστεύσει και οι παράκτε περιοχέ θα βυθιστούν. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απειλή, πρέπει να έχουμε κοινού ε, παγκοσμίου στόχου και η δράση μα να είναι σε τοπικό επίπεδο. Για σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μπορούμε να κερδίσουμε μάχε όπω για την κινητικότητα ή τα κατάλοιπα. Και όταν είσαι πιο κοντά στου πολίτε, είναι πιο εύκολο να του εξηγήσει τη σημασία που έχει η δραστηριότητά τη. Πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα και στην καθημερινή ζωή. Γι' αυτό προτείνω η μάχη κατά τη κλιματική αλλαγή να είναι οριζόντια σε όλου του προπολογισμού για όλα τα ε, δημόσια, του, όλους τους φορείς και η ενέργεια στην οποία, με την οποία θα λειτουργούν είναι 100% ανανεώσιμη και ο κλιματικό αυτό άξονα να του υποβάλει, να μα υποβάλουν και λογαριασμού στην ε, χώρα των Βάσκων από το 2020 θα ε, εφαρμόσουμε αυτή τη βέλτιστη πρακτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενη ομιλήτρια η συνάδελφος κυρία Μέτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, ε, η φροντίδα της γης και του εδάφους μας, όλα αυτά το γνωρίζουμε. Τα Αυτά πρέπει να είναι ο ε, που θα μας βοηθήσει να αποθηκεύσουμε και να δεσμεύσουμε το διοξίδιο του άνθρακα, όλα αυτά ε, όταν δεν γίνονται αυξάνεται η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα στον πλανήτη. Ε, είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι οργανισμοί να έχουν καλή υγεία γιατί ένα μικρό μανιτάρι, ένας μικροοργανισμός ε, μπορεί να ζήσει σε αυτή τη γη μόνο αν εμείς δεν καταστρέψουμε το οικοσύστημά του με χημικά προϊόντα και αν δεν υπερεκμεταλλευτούμε το έδαφος. Έτσι λοιπόν η οικολογική με μετάβαση στη Γεωργία θα μας βοηθήσει να επανεκαθιδρύσουμε ε, την ισορροπία και να δράσουμε κατά της ε, κλιματικής αλλαγής. Ο αέρας, η γη, το νερό είναι θεμελιώδη στοιχεία της ζωής, της βιοποικιλότητας. Ε, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο για την προστασία των εδαφών. Ευχαριστώ επόμενος ο συνάδελφος Πίπερ. Ευχαριστώ. Ε, ε, είναι σημαντικό εμείς ε, να προχωρήσουμε ως πρωτοπόροι με την απαγόρευση των πλαστικών και την ανταλλαγή των εκπομπών. Πρέπει να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες για την κατάργηση των πλαστικών και για το οξυγόνο. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε να σταματήσουμε την καταλήστευση των πόρων στη Λατινική Αμερική, στην Κίνα. Ε, αυτό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες ε, για να μπορέσουμε να τις επηρεάσουμε οικολογικά. Η Πράσινη Συμφωνία δεν έχει να κάνει μόνο ε, με τους ανθρώπους που δουλεύουν στην βιομηχανία του Χάλιβα ή στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχει να κάνει με όλο τον κόσμο δεν έχει να κάνει ε, μόνο με το ότι θα χάσουν κάποια τη θέση τους. Ε, θα πρέπει να προστατέψουμε το περιβάλλον μας, θα πρέπει να εξοικονομήσουμε χρήματα. Ε, η προστασία του περιβάλλοντος είναι και διασκεδαστική. Μια έξυπνη συμφωνία είναι πάντα μια καλή συμφωνία. Ο συνάδελφος Τσαχίν έχει τώρα το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να διεξάγουμε εδώ μια συζήτηση για την οικολογική έκτακτη ανάγκη, την κλιματική έκτακτη ανάγκη, χωρίς να φερόμαστε στα μέτρα τα οποία πρέπει να αναλάβουμε. Γιατί εδώ είναι και τη διαφορά του αν είμαστε πραγματικοί ηγέτε ή αν παριστάνουμε τους ηγέτες στο ζήτημα αυτό. Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι κάνουν πάρα πολλά θετικά πράγματα. Είμαστε όμως πραγματικά οι πιο καθαρή πυρος. Μειώθηκαν σίγουρα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Παρ' όλα αυτά το οικολογικό μα αποτύπωμα, το ανθρακικό μας αποτύπωμα αυξάνεται όλο και περισσότερο φέρουμε εμείς μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Έχουμε πάρα πολλές εισαγωγέ από την Κίνα. Σαφώς θα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις στην κλιματική διπλωματία. Θα πρέπει να καταργήσουμε τις επιδοτήσεις για τα ορεικτά καύσιμα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε πιο φυσικές βιώσιμες λύσεις στα πλαίσια της οικονομίας. Ακούγω την κυρία Φοντερ Λάιν, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τη μείωση του 50% και υπό την ακολουθήσουν και άλλες χώρες θα πάμε στο 55%. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι υποκρινόμαστε ότι είμαστε ηγέτες, δεν συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά υπάρχει κλιματική έκτακτη ανάγκη. Ας είμαστε πραγματικά φιλόδοξοι, εμπράκτος φιλόδοξοι. Η κυρία Κάρλσπρο προέχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το κλίμα και η κλιματική αλλαγή χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα και οι λύσεις βέβαια δεν μπορούν και αυτές να οριοθετηθούν σε σύνορα. Χρειάζεται μια άμεση κλιματική και οικολογική δράση και μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να τροποποιήσουμε τα πράγματα προτού να είναι πάρα πολύ αργά. Νομίζω ότι τα μεμονωμένα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, θα πρέπει να μπορέσουν να κάνουν τις σωστές οικολογικές επιλογές. Αλλά ξέρετε ότι θα μας τυχίσει πάρα πολύ αν δεν λάβουμε τις σωστές αποφάσεις και αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε υψηλά ποσοστά διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήταν θετικό να είχαμε ε, μια κοινή φορολογική βάση όσον αφορά το διοξιδίο του άνθρακα για την κυκλική οικονομία και για τη βιωσιμότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε στο ζήτημα αυτό παντού στον πλανήτη ως Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω επίσης ότι η εμπορική πολιτική που ακολουθούμε θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για την οικονομική μας ανάπτυξη. Μια φύλλο περιβαλλοντική οικολογική ανάπτυξη που θα μας επιτρέψει να ξεφύγουμε από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν το κάνουμε εμείς, ποιο θα το κάνει. Ο κύριος Ένσλι έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ας αποφασίσουμε επιτέλους να βγούμε από τον φαύλο αυτό κύκλο. Η επιστήμη τα λέει ξεκάθαρα τα πράγματα και χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Οι πολιτικοί οι οποίοι δεν ακολουθούν τους επιστήμονες ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ε, στρέφονται κατά τον ίδιο των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο είχαμε 6 εκατομμύρια παιδιά και νέους που διαδήλωσαν τις τελευταίες εβδομάδες στρεφόμενοι κατά των πολιτικών. Όταν έρχονται νέοι και μας ρωτάνε τι κάνετε εσείς που είστε πολιτικός, εγώ για παράδειγμα τους λέω ότι στη δική μου την εκλογική περιφέρεια έχω αναλάβει κάθε δυνατή απόφαση προκειμένου να καταφέρουμε να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030. Ακριβώς αυτό θα πρέπει όμως να κάνουμε όχι μόνο σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο. Ήμουν ένας από αυτούς που κατάφερα να πείσουν τους αξιωματούχους Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν τις επιδοτήσεις διοξιδίου του άνθρακα για την αεροναυτιλία και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει περιοχή και στα άλλα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πράξουν αναλόγως. Αν θέλουμε ένα μέλλον, τώρα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Σας ευχαριστούμε. Γκιούρκ, παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αναφίβολα η κλιματική κατάσταση είναι δεινή και πάρα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό το λόγο συζητήσεις σαν τη σημερινή δεν επαρκούν. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση με τρόπο υπεύθυνο, συντοπιώντας πόσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα. Η βιώσιμη ανάπτυξη επίσης έχει μια πτυχή κοινωνική και μια πτυχή που άπτεται τον ταγωνισμό. Αν επικεντρωθούμε εμεί μόνο στους οικολογικούς παράγοντες, τότε αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε μια οικονομική και κοινωνική έκτακτη ανάγκη και αυτό θα ήταν απαράδεκτο, όσο απαράδεκτη είναι και η ίδια η οικολογική έκτακτη ανάγκη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια οικολογική μετάβαση η οποία να είναι θεμητή από πλευρά ανταγωνισμού. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε μέτρα τα οποία δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση των ενεργειακών τιμών για του πολίτε και δεν θα θέσουν σε καμία περίπτωση ένα αμφιβόλο την οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Α μην δημιουργήσουμε αθέμητε συνθήκε ανταγωνισμού. Α δούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία, όπου καταφέραμε μέσω τη σωστή πολιτική να μειώσουμε τι τιμέ ενέργεια για του πολίτε, προάγοντα παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη. Μπούρκαρτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μα τι άλλο μας μένει παρά να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε σε κατάσταση κλιματικής ανάγκης. Ανεβαίνουν θερμοκρασίες, ε, ε, εξαφανίζονται τα είδη και πολλοί χρειάζεται να καταλήψουν τις αιστείες τους. Αλλά να κηρύξουμε κατάσταση ανάγκης είναι το ένα. Το αποφασιστικό είναι αν ε, θέλουμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, η γεωργική πολιτική πρέπει να στηρίξει τους γεωργούς και τη βιώσιμη γεωργία. Και στις ε, εμπορικές μας συμφωνίες πρέπει να έχουμε δεσμευτικές ρήτρες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά στάνταρ. Πρέπει να έχουμε λοιπόν σαφείς στόχους και συγκεκριμένη εφαρμογή. Αν είμαστε σοβαροί, τότε πρέπει να επενδύσουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον με τη νέα πράσινη συμφωνία για ένα οικολογικό μέλλον. Είναι μόνο η αρχή λοιπόν η κήρυξη της ανάγκη. Μετά πρέπει να κάνουμε και την υπόλοιπη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, εάν η θερμοκρασία της ε, επιφάνειας ε, του πλανήτη αυξηθεί όπως προβλέπεται, θα έχει τρομέρε επιπτώσει. και τα αποτελέσματα της θέρμανσης ε, θα είναι πολύ απτά στην Αρκτική. Η Αρκτική θερμαίνεται με, διπλή, με διπλό ρυθμό από τον υπόλοιπο πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων θα συμβάλλει περισσότερο στην κλιματική αλλαγή. Η ευθύνη για την Αρκτική δεν μπορεί να είναι στα χέρια μόνο των χωρών που είναι γύρω από την Αρκτική. Η μόλυνση στην Αρκτική είναι κυρίως από την Βόρεια Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη. Και η τήξη των πάγων έχει ανοίξει ένα νέο ανταγωνισμό για την περιοχή. Πολλές κυβερνήσεις και εταιρείε θέλουν ε, να αρχίσουν να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς πόρους και να βρουν νέες οδούς ναυσιπλοείας. Και όλα αυτά θα επηρεάσουν ε, την ασφάλεια στην Ευρώπη και ευρύτερα. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη των Παρισιών, πρέπει να μειώσουμε τάχιστα τις εκπομπές και πρέπει να προετοιμαστούμε για τις αλλαγέ που θα προκύψουν για να αποφύγουμε τις εντάσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δουμπερνάι Κλουνενμπέρκ. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν ε, οι περισσότεροι πολίτες τι συμβαίνει στον πλανήτη. Δεν καταλαβαίνουμε τι θα γίνει, τι επιπτώσεις θα έχουν οι ενέργειές μας. Θα είναι παγκόσμιες και πολύ ε, σοβαρές για πολύ μετά την ε, δική μας ζωή. Δηλαδή μόνο όταν δούμε πόσο άθλια είναι η κατάσταση, όταν θα την έχουμε στο κεφάλι μας, όταν θα την μυρίζουμε, όταν την αισθανόμαστε στο πετσί μα, τότε μόνο θα δράσουμε. Πρέπει να γίνει μια βαθύτερη αλλαγή νοοτροπία. Όλοι μα και οι κοινωνίε πρέπει να μαθαίνουμε κάθε μέρα. Να παίρνουμε τι σωστέ αποφάσει που θα διατηρήσουν τη ζωή. Για παράδειγμα, τι κουλτούρα κινητικότητα έχουμε. Κατανάλωση. Τροφίμων. Πώ θα καθορίσουμε την ευημερία μα. Τι σημαίνει ευημερία. Και φυσικά πρέπει να ληφθούν συλλογικέ αποφάσει. Μέτρα για την αγορά και για τις τεχνολογίες. Χρειαζόμαστε όλοι λοιπόν από κοινού με τους επιστήμονες, τους πολιτικούς, τους φιλοσόφους και τους ε, καλλιτέχνες να δράσουμε. Με μια θετική δράση, με μια, ένα θετικό όραμα, να δείξουμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Αν υπάρξει αυτή η αλλαγή κουλτούρας θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο για να προστατεύσουμε το κλίμα μας και την βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μπέντελε. Εφόσον καλούμε την κατάσταση επίγουσα, τότε πρέπει ε, να υπάρξει περισσότερη ε, εξουσία στην εκτελεστική ε, εξουσία και θα παραβλέψουμε κάποια θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οι βουλευτές από τα μεγάλα κράτη ξέρουν ότι στο μέλλον όλες, όλα τα μέτρα θα έχουν ως κριτήριο ε, αν θα επιτρέψουν καθαρότερο περιβάλλον και περισσότερη υγεία. Στις πόλεις όπως το Βερολίνο, το Παρίσι, στη Τζακάρτα, στην πόλη του Μεξικού ή το Πεκίνο έχουμε όλο και περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω του πληθυσμού, των μεταφορών κτλ. Όμως ε, έχουμε και περισσότερη τεχνογνωσία τώρα. Έχουμε τεχνολογίες που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα. Έκκληση προς την Κομισιόν ιδιαίτερα να δούμε τι δυνατότητες έχουν οι πόλεις για να αντιδράσουν, ούτω ώστε να αναδιαμορφώσουμε τις πόλεις μας για να σώσουμε το περιβάλλον μας. Ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Περέιρα. Κυρία Πρόεδρε, Μερικές φορές πρέπει να εξηγούμε για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε κάτι, όχι πάντως σήμερα. Σήμερα οι επιχειρήσεις μας, οι πόλεις μας, οι πολίτες